Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που προεδρεύω για λίγο χρονικό διάστημα αυτή την ε, συνεδρία της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Βέβαια το πρόγραμμα είναι η συγκρότηση όλων του Προεδρείου της Επιτροπής αυτής με εκλογή Προέδρου και κατόπιν και Αντιπροέδρων. Απαρτία φαντάζομαι υπάρχει. Κανένα πρόβλημα, δεν βλέπω, είναι πλήρης η αίθουσα. Όλοι χαίρονται που ξαναβρίσκονται εδώ. Λοιπόν, μία απλή ερώτηση. Οι υποψηφιότητε για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής αυτής. Ο κύριος Δικάστρο, ρωτώ τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, είναι υποψήφιος. Ναι, ο κύριος Δικάστρο, ναι, γνέφει καταφατικά. Είναι υποψήφιος πράγματι. Κατά δεύτερον, θέλω να ξέρω εάν υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι για το αξίωμα αυτό. Donc il n'y a qu'un seul candidat, c'est M. υπάρχει, ο κύριος Δικάστρο. Βλέπω ότι συμπλήρωσε την δήλωσή του οικονομικών συμφερόντων. Είναι πολύ εντάξει λοιπόν και γι' αυτό σας προτείνω να περάσουμε στην εκλογή του διαβοής, εκτός αν διαφωνεί κάποιος και θέλει καλύτερα μυστική ψηφοφορία. Δεν βλέπω. Λοιπόν, προτείνω να εκλέξουμε διαβοή στον κύριο je vais donc lui céder la place. Euh, Θα τον καλέσω λοιπόν να ανελάβει εδώ τον θόκο του Προέδρου. Το παραδίδω με μεγάλη ευχαρίστηση. Και τώρα εκείνος πρέπει να δουλέψει. Bene, grazie della fiducia. Diamo subito inizio alla procedura di... ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής των αντιπροέδρων. Εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Με πληροφορούν ότι η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όρισε τον κύριο Νιτσελέσκου ως πρώτο αντιπρόεδρο. Κύριε Νιτσελέσκου, δέχεστε αυτή, την ε, πρόταση. Δέχομαι. Ξέρω ότι ο κύριος Νιτσελέσκου έχει κάνει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Ρωτώ, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. ουδής. Τότε κηρύσω τον κύριο Νισελέσκο πρώτο αντιπρόεδρό μας. Σας παρακαλώ κύριε Νισελέσκο, ελάτε δίπλα μου. Α Ας έρθουμε στην εκλογή του δευτέρου αντιπρόεδρου. Με πληροφορούν ότι η ομάδα των Παρσίνων όρισε τον κύριο Μποβέ ως δεύτερο αντιπρόεδρο. Κύριε Μποβέ, δέχεστε αυτή την πρόταση? Ναι. Ξέρω ότι ο κύριος, βλέπω ότι ο κύριος Μποβέ έχει κάνει τη δήλωση οικονομικών προσωπικών συμφερόντων. Ερωτώ, υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για τη δεύτερη αντιπροεδρία? ουδής. Άρα ο κύριος Μποβέ είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Και τον παρακαλώ να έρθει να καθίσει δίπλα στον κύριο Νικολέσκο. Για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Με πληροφορεί η γραμματεία ότι η ομάδα SCR όρισε τον κύριο Μπατσακόσκι ως τρίτο αντιπρόεδρο. Κύριε Μπατσακόσκι, δέχεστε αυτή την πρόταση? Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας, Μπατσιακόσκι. Ξέρω ότι ο κύριος Μπατσακόσκι έχει κάνει δήλωση προσωπικών οικονομικών συμφερόντων Ερωτώ, υπάρχει άλλος υποψήφιος για την τρίτη αντιπροεδρία? Ουδής. Τότε ο κ. Μπασιόφσκι ορίζεται ως τρίτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, ελάτε στο βήμα. Δίπλα στον κύριο Μποβέ. Και τέλος, εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου, του τετάρτου συγγνώμη αντιπροέδρου, η ομάδα Άλντε των Φιλελευθέρων όρισε τον κύριο Πόλσον ως τέταρτο αντιπρόεδρο. Κύριε Πόλσον, δέχεστε αυτή την πρόταση. Ξέρω ότι έχει κάνει τη δήλωση προσωπικών συμφερόντων ο κ. Πόλσον. Υπάρχει άλλος υποψήφιος για τη θέση του τετάρτου αντιπρόεδρου. Όχι. τότε ο συνάδελφος Πόλσεν, τέταρτος αντιπρόεδρος και καλείται να καθίσει δίπλα στον συνάδελφο Βασιβόφσκι. Έτσι συνεσήφθη το Προεδρείο της Επιτροπής μας. Πριν κλείσει η συνεδρίαση, θα ήθελα να σας πω μερικές πολύ σύντομες σκέψεις. αγαπητοί συνάδελφοι. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω με την σύμφωνη γνώμη σας στην Προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Με τιμά η εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου και σας διαβεβαιώνω ότι η δέσμευσή μου ως Προέδρου θα είναι η μέγιστη δυνατή προκειμένου να παίξουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στα στοιχεία και ενδείξεις που θα φύγουν από το όργανο αυτό εδώ προς τα έξω προκειμένου να λαμβάνει σωστές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Το σύστημα της συναπόφασης σωστά τονίζει τις εξουσίες του Ευρωκοινοβουλίου αποδίδοντας επιτέλους στο σοβαρό αυτό θεσμό και σε αυτούς που εξελέγησαν από τους Ευρωπαίους πολίτες ένα πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με προνόμια που μέχρι χθε αποκλειστικά τα είχε το Συμβούλιο. Αν τα επιτρέψει φυσικά αυτά το Ιρλανδικό Δημοψήφισμα. Σήμερα η δημιουργία των νέων βασικών επιλογών γίνεται με ένα μηχανισμό όπου ενισχυμένος είναι ο ρόλος του εκλεγμένου Ευρωκοινοβουλίου. Κατά συνέπεια είναι πιο άμεσος και ισχυρός ο ρόλος και για τις αποφάσεις εκ μέρους των συναδέλφων που κάθονται στα έδρανα εδώ, με δημοκρατικές αποφάσεις που έχουν πάρει οι εκλογείς και οι πολίτες της Ευρώπης μας. Αυτό επίσης είναι σημαντικό όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, που είναι κοινή κληρονομιά όλων των πολιτών. Μια νέα δομή λοιπόν στη σύνθεση και στη λήψη των αποφάσεων και στις επιλογές και τις αρμοδιότητες όσον αφορά την υγειορική πολιτική. Θα είναι η προσωπική μου δέσμευση όλα αυτά να τα προσπίσω, να τα υπερασπίσω, να τα ενισχύσω και τυπικά και κυρίως συγκεκριμένα. Και όλα αυτά σε ένα κοινοβούλιο που καλείται να οικοδομήσει την Ευρώπη του μέλλοντος. Είναι ο καιρός των επιλογών. Οι αποφάσεις που θα πάρουμε σε αυτή την πενταετία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Εμείς θα δώσουμε ουσία στις κατευθύνσεις και στους πόρους της κοινή γεωρικής πολιτικής μετά το 2013. Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει και εμείς αγαπητοί συνάδελφοι καλούμαστε να παίξουμε έναν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για να καθοδηγήσουμε προς μια συζήτηση που θα υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της Ευρώπης προκειμένου να υπάρχει ένας κοινωνικός και οικονομικός ορίζοντας σύγχρονος και βιώσιμος. Για μένα είναι τιμή να εκπροσωπώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας τις εργασίες που είμαι σίγουρος ότι θα εκπονήσουμε με ευθύνη και με συμμετοχή όλων σας. Σας ευχαριστώ και πάλι και